Friends we'll start the meeting. Uh, it's past... Να ξεκινήσουμε αγαπητοί συναδελφοί τη συνεδρίασή μας. Είναι 9 και 10. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Αλλά φαντάζομαι ότι όσοι είστε εδώ θα κάνετε πολύ σκληρές ερωτήσεις στον Επίτροπο. Αφού μας κάνει την εισαγωγή του. Όπως ξέρετε αυτό είναι ένα κομμάτι του διαρθρωμένου διαλόγου. Είχαμε τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης και τον Επιτροπό Τάισεν εδώ στις αρχές του Μάη και τώρα καλωσορίζουμε τον Επίτροπο Γυρκή Κατάινεν. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη Ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι στη συναδρίαση της Επιτροπής σας. Και βεβαίως θα χαρώ πολύ να ακούσω και τις απόψεις σας για διάφορα θέματα και προτεραιότητες που έχουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας δύο πράγματα για τη διαδικασία της Λευκής Βίβλου. Αυτό που λέω συνήθως όταν επισκέπτομαι κράτη-μέλη και στους ε, ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και στους κυβερνήσεις είναι ότι είναι σημαντικό να ε, καταλάβουμε ότι μόλις αποχωρήσει η ε, το Ηνωμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα Ευρώπη των 27. Και αυτή η νέα Ευρώπη δεν θα είναι όπως η παλιά, θα είναι μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο θα βρεθούμε σε μια φάση της διαδικασίας όπου πολλοί τομείς της ε, πολιτικής θα προχωρήσουν. Η κοινωνική διάσταση, η άμυνα, το EMU θα είναι από τους τομείς που θα περιμένουμε πολλές προτάσεις από τα κράτη-μέλη και από τις πολιτικές ομάδες και είμαστε στα μέσα μιας δυναμικής, μιας ζωντανής διαδικασίας και αυτό νομίζω ότι θα ενεργοποιήσει τα κράτη-μέλη. Πριν από λίγους μήνες βρισκόμασταν σε μια υπαρξιακή κρίση, μάλλον εν το μέσο πολλών υπαρξιακών κρίσεων. Άνθρωποι που δουλεύουν και ασχολούνται με το μέλλον της Ευρώπης, ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ήμασταν όλοι σε φάση διαχείρισης της κρίσης, να δούμε πώς μπορούμε να διασώσουμε όσα έχουμε. Πολλοί μπορεί να σκέφτηκαν ότι ίσως αυτή να είναι και η αρχή του τέλους αλλά δεν φαίνεται να έχει γίνει αυτό. Και επίσης έχουμε και διάφορες εξωτερικές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν την δική μας εξωτερική κατάσταση. δική μου βέβαια προσωπική άποψη είναι ότι μάλλον μας φέρνουν πιο κοντά αυτές οι εξωτερικές κρίσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν ο κόσμος είναι ε, τόσο περίεργος όπως είναι τώρα, ίσως είναι καλύτερο να έρθουμε πιο κοντά, να είμαστε κοντά όλοι εμείς που πιστεύουμε στο κοινωνικό κράτος, ε, στην, που θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, μια, ένα καλύτερο κόσμο μέσα στην παγκοσμιοποίηση, που θέλουμε να παρουσιάσουμε τις αξίες και όχι μόνο τα συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια πολιτική δύναμη στον κόσμο που να μπορεί κανείς να την εμπιστευτεί. Και μάλιστα ήταν πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε όλες αυτές τις ε, αντιπροσωπείες ε, και ε, σε ταξίδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλές χώρες του κόσμου, χώρες από την Ασία ή τον Κόλπο, την Νότια Αμερική. Φαίνεται να πιστεύουν ότι τώρα πρέπει να ενδυναμώσουν και αυτές τις σχέσεις τους με τις με την Ευρώπη, γιατί πιστεύουν αυτό που πιστεύουμε κι εμεί για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφωνίε και επί τη ουσία σημαντικέ διαφωνίε μερικέ φορές, υπάρχουν κάποιοι τομείς που διαπερνούν τις πολιτικές γραμμές και πρέπει να δούμε το μέλλον. Εγώ χαίρομαι που κινούμεθα γρήγορα από την, και περνάμε από την υπαρξιακή κρίση σε μια κατάσταση όπου οραματιζόμαστε το μέλλον της Ευρώπης. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης. Τι περιμένουμε. Πρέπει να εμφαρίνουμε τους πολίτες να μας πούνε τι περιμένουν από την Ευρώπη δεν χρειάζεται να ξέρουν κατά ανάγκη τις διαφορέ μεταξύ των θεσμικών οργάνων. αυτό μπορεί να είναι λίγο περίπλοκο κάποιες φορές, αλλά το βασικό είναι να ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια και τους πολίτες των κρατών μελών να μας πούν τι περιμένουν από το μέλλον της Ευρώπης. Περιμένουν περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, τι περιμένουν. Γνωρίζετε λοιπόν ότι Έχουμε δημοσιεύσει τη Λευκή Πίβλο και κάποια έγγραφα προς ε, διαβούλευση. Και θα ήθελα να τονίσω ότι ο έγγραφο που ασχολείται με την ενίσχυση της ε, παγκοσμιοποίησης που τονίζει πώς ε, θα, από την πλευρά της Κομισιόν πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση καθώς επίσης και ένα έγγραφο για την κοινωνική διάσταση των πραγμάτων. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν και οι τεχνολογικές αλλαγές αλλάζουν τη ζωή μας και κάποιοι, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και αλλού, είναι, ε, μπορεί να μπουν στον ε, πειρασμό να περιχαρακωθούν στα εθνικά του ε, σύνορα. Αυτή η διαδικασία όμω δεν μπορεί να ανατραπεί, δεν μπορεί να αντιστραφεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να δώσει μια μορφή στον, στην παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με τα δικά τη συμφέροντα και τι αξίε. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιώντα τα μέσα που έχουμε, ανοίγοντα τι αγορέ και προωθώντας την τεχνολογική πρόοδο για να προωθήσουμε του στόχου μα να προωθήσουμε τα δικαιώματα και την ανθρώπινη ευημερία. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια πηγή άγχους για πολλούς πολίτες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε τα στοιχεία αυτά και να δούμε πού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι πολίτες συνεχίζουν να υποφελούνται από την παγκοσμιοποίηση. Οι πολίτες μπορούν να σπουδάσουν, να ζήσουν, να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες, έχουν επαφές ε, μέσω, των, ε, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του ίντερνετ, αντιμετωπίζουν, ε, ανταλλάσσουν απόψεις, βλέπουν νέες κουλτούρες και πολιτισμούς. Οι φοιτητές μπορούν και online να σπουδάσουν, μπορούν να φοιτήσουν σε ξένα πανεπιστήμια οι χώρες μπορούν να παράξουν περισσότερα με λιγότερα, με, εξειδίκευση, με αυτό που κάνουν καλύτερα και χρημα, ε, εκμεταλλευόμενες τις ε, ε, οικονομίες, αγοράς, οικονομίες κλίμακας. Ε, υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές, ε, πολίτες παντού ζητούν υψηλότερη ποιότητα προϊόντα και υπηρεσίες. Και όχι μόνο οι μεγάλες εταιρείε φαλούνται από αυτό, αλλά και οι μικρομεσαίες. 80% των εξαγωγέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάθε ένα δις ευρώ εξαγωγών υποστηρίζει 14.000 θέσεις εργασίας. Και είναι αλήθεια ότι αυτά τα ωφέλη δεν είναι καταναμημένα ε, εξίσου στην, ε, στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες και μεταξύ των πολιτών μας. Το κόστος ε, το, είναι τοπικό πολλές φορές και κάποιες περιφέρειες επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τις άλλες. Οι ανάγκες για εργατικό δυναμικό με υψηλά προσόντα προωθεί την τη δημιουργία προβλημάτων για άτομα που δεν έχουν τόσο πολλά, τόσο πολλές δεξιότητες. Είναι σημαντικό όμω να πούμε ότι η παγκοσμιοποίηση από μόνη τη δεν δημιουργεί νικητέ και ιτημένου, αλλά τα αποτελέσματά τη έχουν να κάνουν με το πώ διαρθρώνεται. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρώπη να δώσει μια κατεύθυνση στην παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να γράψουμε τους κανόνες, να διαρθρώσουμε την ε, παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με τις αρχές μας, ας πούμε όταν μιλούμε για, τον, για το ε, εμπόριο που θα βασίζεται σε κανόνες. Το να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ε, περιφερειών που έχουν πολλά πλεονεκτήματα και όχι, ουσιαστικά κρατά τους πολίτες φυλακισμένους. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό και να κινηθούμε έξυπνα εκεί που χρειάζεται. Είναι σημαντικό να, είμαστε, να μιλούμε με μία φωνή έτσι ώστε οι κοινωνίες μας να είναι πιο ανθεκτικές. Καταρχάς υπάρχει ε, η πτυχή της ε, οικονομίας που πρέπει να κοιτά προς τα έξω. Πρέπει οι οικονομίες μας να είναι πιο ανταγωνιστικές προς τις παγκόσμιες αγορές, γιατί αυτή είναι η βάση για να υπάρχουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και ευημερία. Η ανθεκτικότητα όμως έχει και μια εσωτερική διάσταση όταν πρόκειται για τους πολίτες μας και για τις κοινωνίες μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περαιτέρω επενδύσεις στην εκπαίδευση και στις ε, δεξιότητες. Η διαβίου μάθηση επίσης είναι ένα σημείο κλειδί. Η πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας είναι ένας τρόπος επίσης για να αναδιανύμουμε τον πλούτο στην κοινωνία και να προωθήσουμε τις τέσσερα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους. Εφόσον υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα της ε, εκπαίδευσης και κυρίως ό,τι αφορά την κατάρτιση των ε, ε, εκπαιδευτικών δεν κάνουμε τελικώς αρκετά από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε δίκαιες κοινωνίες και βιώσιμες κοινωνίες με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό θέλω να το τονίσω. Κυρίως την ποιότητα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Και πάμε τώρα στο θέμα των δεξιοτήτων. Όπως ξέρετε, Πέρσι ξεκίνησε ένα νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες στην Ευρώπη, ζητώντα από τις περιφέρειες, τις ε, τοπικές αρχές, τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρου, του ε, τους εργαζόμενους, εργοδότε, εργοδότες, την κοινωνία των πολιτών, να συνεργαστούν για να βελτιώσουν τις δεξιότητες στην Ευρώπη και να αντιμετωπίσουν τι ε, μεγάλε αλλαγέ τη κοινωνία. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα έχουν τις σωστές δεξιότητες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ε, δραστικές και πολλές φορές μη αναμενόμενες αλλαγές στην κοινωνία μας δεν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζεται κανείς να έχει για να είναι καλός επιχειρηματίας ή για να μπορεί να κρατήσει τη θέση εργασίας, τους, εργασίας του και αυτών που, πρέπει να είναι, που χρειάζεται κανείς για να είναι σωστός πολίτης και ενσωματωμένος στην κοινωνία που ζει. Στο πλαίσιο της, ε, του θεματολογίου για τις δεξιότητες, η Κομισιόν ήδη έχει κάνει πολλές προτάσεις για να βελτιώσει ας πούμε, την ποιότητα των, της δημιουργίας των ε, δεξιοτήτων ή την ορατότητα και τη συγκρισιμότητα αυτών. Μετά, θα ήθελα να στραφώ στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Μαζί και με το έγγραφο ε, διαβούλευσης για, για την κοινωνική διάσταση έχουμε υιοθετήσει και τον πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Οι θεμελιώδεις αρχές είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να, έχει κοινωνική, να, να επιφέρει κοινωνική πρόοδο και αυτό αποτέλεσε τον ακρογωνίο λίθο της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινωνικό μας μοντέλο είναι επιτυχές. Η Ευρώπη έχει, τις, ε, πιο, ε, έχει την ε, πιο ισότιμη σε εισαγωγικά κοινωνία του κόσμου. Το κενό της απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει μειωθεί κατά 30% και επίσης ε, προχωρούμε ε, ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερες ε, θέσεις εργασίας με 232 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αυτό είναι το υψηλότερο στοιχείο αριθμητικό που είχαμε ποτέ. Έχουμε βεβαίω δραστική ψηφιοποίηση και γύρανση των κοινωνιών μας. Αν αυτά τα θέματα δεν τα αντιμετωπίσουμε, μπορεί να απειλήσουν τη βιωσιμότητα του κοινωνικού μοντέλου μας και να επιτείνουν ακόμη περισσότερο τις ανισότητες. Ο Ευρωπαϊκό Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων ε, αποτελεί μια επεξίδα για τη βελτίωση τη απασχολησιμότητα και των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και ε, νομίζω ότι ε, μπορεί να επιτύχει το σκοπό τη αντιμετώπισης τη παγκοσμιοποίηση. Καλύτερη διανομή των επιδομάτων σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή του και με την κοινωνική προστασία θα βοηθήσει του πολίτε να βρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασία και να μπορούν να αντέξουν τι αλλαγέ οι επικεντρωμένες ε, στοχευμένες επενδύσεις στην κοινωνική ε, ενσωμάτωση ε, ανάτομων όπως οι μετανάστες θα βοηθήσουν να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Τώρα λοιπόν είναι η σειρά των κρατών μελών να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή και να αποφασίσουν πώς θέλουν να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οι πολιτικές που εξασφαλίζουν ε, ωφέλη για όλους σημαίνει ότι θα πρέπει να, έχουν, να τύχουν και σημαντικών επενδύσεων. Κάτι που μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο μέσω μιας ε, ανθούσας οικονομίας. Γι' αυτό πρέπει, φαίνεται, γιατί πρέπει να προωθήσουμε την κοινωνική πρόοδο. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα συνεχίσει να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο έτσι ώστε οι αρχές του πυλώνα να μπορούν να μεταφραστούν σε πράξεις. Αυτό βεβαίω θα βασιστεί στο ήδη στεναρό κοινωνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και βεβαίως η κοινωνική πτυχή πάντα ενισχύεται. Να πω δύο λόγια τελειώνοντας για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι ε, συστάσει αναχώρα αυτή τη χρονιά ε, επικεντρώνονται κυρίω στην ενσωμάτωση, στην ένταξη. Οι ανισότητε δεν μα χωρίζουν, ε, δεν χωρίζουν απλώ τι κοινωνίε μα, αλλά φρενάρουν και την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική μα ανάπτυξη. Η δημιουργία θέσεων απασχόληση μέσω συνδυασμού τη αγορά-εργασία και της οικονομικής μεταρρύθμισης μπορούν να βοηθήσουν και ως προς αυτό οι επενδύσεις είναι σημαντικές. Πρέπει να έχουμε καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας και αυτός θα είναι ο στόχος μας για το μέλλον. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων αλλά και η ετροποποίηση αυτών ο, μεγάλο, ο ταχύς ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών επιβάλλουν την βελτίωση στην ε, πρόσβαση της ε, ε, εκπαίδευσης και της επαγγελματική κατάρτισης αλλά και της διαβίου μάθησης. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης των πολιτών και δίνουν στις επιχειρήσεις ένα καλό, με σωστές δεξιότητες, εργατικό δυναμικό. Η προώθηση της ε, ε, ενεργού ε, επαγγελματικής ζωής μπορεί να αντιμετωπίσει την ε, πίεση που δέχονται τα συστήματα κοινωνικής ε, ασφάλισης. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν ε, μεταρρυθμίσεις και στις πολιτικές για την υγεία και την εργασία έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Η μείωση της φτώχειας και η αντιμετώπιση κάποιων ανισοτήτων σε ό,τι αφορά τους μισθούς τα εισοδήματα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της επάρκειας και της κάλυψης του ελέγχου του εισοδήματος ή των προγραμμάτων επιδοτήσεων. Επίσης αυτό μπορεί να γίνει μέσω της αντιμετώπισης των ανισοτήτων σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες και τη καλύτερη πρόσβαση σε υψηλή ποιότητα, κατάρτιση και εκπαίδευση, καλύτερη στέγαση, υγεία. Το πήραμε με, τις, ε, με το βασικό εισόδημα ξεκίνησε και στη Φιλανδία το 2015 ε, προσπαθώντας να βρούμε τρόπους να αναδομήσουμε το σύστημα κοινωνική ασφάλισης και να απαντήσουμε στι αλλαγέ στην ε, αγορά εργασία. Και το πείραμα αυτό διαρευνά το πώ μπορεί το σύστημα να ενισχυθεί για του δικαιούχου αυτών των επιδομάτων και πώ μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό έτσι ώστε να δώσει κίνητρα στην, ε, για την εργασία ανάλογα με τι συστάσει αναχώρα βεβαίω και ό,τι αφορά τη δική μα χώρα, τη Φιλανδία. Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από, ένα, από μια πολύ περίεργη διάδραση μεταξύ διαφόρων ειδών επιδομάτων κάτι που καταλήγει σε κενά εισοδηματικά σε σχέση με κάποιες ε, κοινωνικές ομάδες. Η μελέτη λοιπόν που έχει γίνει θα βοηθήσει να, να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το πρόγραμμα και ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να έχει στην ε, συμπεριφορά ε, των εργαζομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κυρίες και κύριοι παραμένει δεσμευμένη στην κινητικότητα των εργαζομένων, στην κοινωνική προστασία και τώρα είναι η σειρά των κρατών μελών να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή. Αν θέλουμε όντω οι κοινωνίε μα να ανθίσουν και να ευημερούν σε, μια, σε ένα ψηφιοποιημένο κόσμο, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και πρέπει βεβαίω να έχουμε και ανθεκτικέ κοινωνίε. Αυτά και σα ευχαριστώ. Thank you for that. Ευχαριστούμε για αυτήν την συζήτηση. Έχουμε κάμποσους συντονιστές εδώ αλλά θα ξεκινήσω ακόμη και αν κάποιοι λείπουν. Ε, δύο λεπτά για τον καθένα σας. Ο κύριος Μπέκερ και μετά ο κύριος ε, Τσαμπών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Ε, και Ευρωπαίοι πολίτες. Ελπίζουμε να είστε πολύ άριθμοι, καθώς έχουμε και τις οθόνες εδώ για τη μετάδοση στο διαδίκτυο, στη συζήτηση μα με τον κύριο Κατάινεν. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε και για την εξομολόγησή σας ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε μια Ευρώπη των 27 πλέον. Αυτό είναι το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, ήταν πολύ σαφή η δήλωσή σας και εδώ συμπεριλαμβάνουμε την κοινωνική Ευρώπη, αυτό είναι που μας αφορά. Ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλουμε να είναι αυτό η ραχοκοκαλιά της επικουρικότητας των ε, κρατών μελών. Και αυτό είναι ε, και αυτό που κατανοούμε εμεί για πολλού τομεί τη κοινωνική πολιτική, στου οποίου θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο μέλλον. Πολύ σωστά τονίζεται και τη διάσταση τη παγκοσμιοποίηση. Η Ευρώπη πρέπει να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητά τη από τη μια και από την άλλη, όπω λέτε, να αναλάβει ηγετικό ρόλο ω κοινωνική επίση ένωση. Αυτό ε, επιδιώκουμε. Η εκπαίδευση, οι δεξιότητε, τα προσόντα για ε, υψηλότερο επίπεδο απασχολησιμότητα Αυτά είναι λύσεις για να έχουν περισσότερη απασχόληση οι πολίτες, ιδίως οι νέοι συμπεριλαμβανομένων και πολύ χαίρομαι που το άκουσα, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, των δασκάλων. Αυτό είναι το κλειδί για το μέλλον. Έχω λοιπόν τρεις ερωτήσεις και ελπίζω να μπορέσω να είμαι σύντομος. Τα απορίσματα στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την εγγύηση των νέων δείχνουν ότι περίπου ότι μάλλον δεν υπάρχουν πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι η αιτία είναι ότι δεν ήταν πολύ φιλόδοξε οι κυβερνήσει των κρατών μελών. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε και είναι ένα σοβαρό εγχείρημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τη δουλειά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τίποτε ιδέε, όχι μόνο για το πώ να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για να την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων, αλλά για να βελτιώσει και την λειτουργία αυτής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Με άλλα λόγια, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο είδος, κάποιο κίνητρο που μπορούμε να προσφέρουμε για να το πω έτσι, ε, κίνητρο που να ασκήσει όμως πίεση στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τον ε, μεταβαλλόμενο κόσμο γύρω μας και ήδη σε ψηφιακό επίπεδο τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα από σήμερα. Δεν μιλάμε για κάποιο μακρινό ορίζοντα για το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένου πολιτικούς στόχους και μέτρα. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την Επιτροπή προς αυτήν την ε, κατεύθυνση για να αντιμετωπίσει τις ε, σημερινέ εξελίξεις με λύσεις που να είναι κατάλληλες για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε τίποτα ιδέε ήδη. Και πώς διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα για αυτές, αν τις έχετε. Η ψηφιοποίηση και αγορά εργασία δηλαδή, με τα κοινωνικά θέματα ταυτόχρονα, πώς συνδυάζονται. Και το τρίτο που θέλω να πω αφορά τον, κοινωνικό, τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πολύ σημαντική ε, προσπάθεια, την καλωσορίζω θερμά. Και υπάρχουν 20 αρχές και μια νομοθετική πρόταση για την εξισορρόπηση επαγγελματικού ιδιωτικού βίου. Η ερώτηση είναι τι νομικό καθεστώς μπορεί να επιτύχει αυτός ο πυλώνας, τι νομικό καθεστώς έχει και τι μπορούμε να περιμένουμε, τι να ελπίζουμε. τι προθέσεις υπάρχουν. Έχετε τίποτε συγκεκριμένες ιδέες για το τι να περιμένουμε και θέλω να ολοκληρώσω εκφράζοντας την ε, πλήρη ικανοποίησή μου για την ποιότητα της συνεργασίας που έχουμε και την ποιότητα του διαλόγου μας με την Επίτροπο Τάισον. Πρέπει να υποθεί πολύ ξεκάθαρα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κυρία Στάινρουκ. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, για τα όσα μας είπατε. Χρειάζεστε μια, χρειαζόμαστε μια πολιτική δύναμη που μπορούμε να εμπιστευόμαστε. Είπατε και εντός και εκτός και το συμμερίζουμε απολύτως. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χώρα πέρασε την κρίση αυτή και είναι και επιτυχής αλλά αυτές οι χώρες που ήταν πιο επιτυχίε ήταν αυτές που είχαν πιο ισχυρό κοινωνικό κράτος. Δεν υπάρχουν λοιπόν αντιφάσεις εδώ, το ένα δεν εξαιρεί το άλλο, η ευελιξία και η ασφάλεια πάνε χέρι-χέρι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ιδέα της εσωτερική αγοράς, η οποία πάντα θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε. Έχουμε ελευθερίε που είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικέ, αλλά ταυτοχρόνω σε πολύ σημαντικούς τομείς, κοινωνική ασφάλιση, φορολογική πολιτική και σε πολλούς άλλους τομείς βέβαια, έχουμε κατακαιρματισμένα εθνικά συστήματα και αυτό βεβαίως δεν διευκολύνει τα πράγματα. Και ακριβώς τώρα βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη όπου οι ανισότητες δυστυχώς δεν μειώνονται αλλά αυξάνονται. Οπότε είναι απολύτως απαραίτητο εκείνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να δραστηριοποιηθεί. Οπότε πραγματικά να έχετε μεγάλες προσδοκίες για, σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό α, πυλώνα. Είπατε για τις διαφορές ε, των αντρών και των γυναικών. Οι διαφορές ε, μειώνονται. Δεν θα ήταν καλό Ούτω ή άλλω δεν συγκρίνουμε τα δεδομένα του 1960, μιλάμε για το 2017 και πραγματικά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα ώστε να μπορέσει να μειώσει αυτέ τι αλλαγέ, τι διαφορέ και υπάρχουν και πολλά σε ό,τι αφορά τι νομοθετικέ πράξει που μπορούν να προωθηθούν. Ας πούμε η οδηγία για την αντιμετώπιση των, ε, της διακριτικής μεταχείρισης που έχει χρόνια που είναι παγωμένη. Δεν πρέπει κάτι να γίνει από αυτού. Ε, άλλο σημείο. Οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Περιμένουμε ένα νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Και βλέπουμε όλο και περισσότερο οι πολίτες να, να ξεφεύγουν από, τα, από τις κοινωνικές ε, δυνατότητες. Ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπιστεί η ε, φτώχεια με την σχετική στρατηγική κατά της φτώχειας. Υπάρχει η εγγύηση για τους νέους και επίσης πρέπει να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας οι οποίες όμως θα έχουν ε, βασικά έναν πυρήνα κοινωνικής προστασίας κάτι που δεν θα είναι απλώ μια υποσημείωση σε ένα νομοθετικό κείμενο, αλλά που θα μπορεί να αλλάξει την κατάσταση των πολιτών. Και ένα ερώτημα για σας. Με την κοινωνική ασφάλιση τι γίνεται. Βλέπουμε ότι έχουμε την, ε, για την ε, πρόταση για την, ε, για την κάρτα για, τις, τα κοινωνικά θέματα, έχουμε την, τις σχετικές οδηγίες, Υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο διάφορα α, στοιχεία για την υποβολή αυτής της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης. Και εδώ πρέπει να έχετε πάλι μεγάλες ε, προσδοκίες. Ξέρουμε ότι αυτό βέβαια είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας, αλλά εδώ η ε, αφοσίωση σε το θέμα αυτό της Κομισιόν είναι απαραίτητη. Υπάρχει και ψηφιακή ατζέντα. Γιατί να μην έχουμε μια ψηφιακή κάρτα ασφάλισης ας πούμε και κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να με ένα κλικ να αποδείξει ποιο είναι και αν μπορεί όντω, αν είναι επιλέξιμος για κοινωνική ασφάλιση ή επιδόματα. Έχουμε επίση πολλά ε, κενά σε ό,τι αφορά του ελέγχου. Οπότε εσεί τι σχέδια έχετε. Μας ε, είπατε πολύ ωραία γενικά πράγματα, αλλά τώρα ακριβώ λόγω και το ότι τελειώνει η θητεία είναι σημαντικό να παρέμβουμε για να έχουμε πραγματικά προστιθέμενη αξία για τους πολίτες. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε ο κύριος Τσαμπών. Καλημέρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σχολιάσω ένα-δυο σημεία που ε, μας αναπτύξατε και εσείς σήμερα το πρωί. Μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες είναι να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Αυτό είναι μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Και αυτοί που έχουν ερωτηθεί ε, αν έχουμε κάνει αρκετά για την περίπτωσή του. είναι βεβαίως οι ίδιοι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτού πρέπει να έχουμε κατά νου. Πρέπει να παραμείνει μια πρώτη μας προτεραιότητα αυτό γιατί οι νέοι είναι το μέλλον της Ευρώπης. Είναι η πραγματικότητα αυτή και είναι κάτι το λογικό. Ε, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αντιμετωπίζουμε την ανεργία των νέων. Όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε, ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την εκπαίδευση συγκεκριμένα και την ε, διαβίωμα την επαγγελματική κατάρτιση μάλλον. Θα πρέπει να καταβάλουμε πολύ περισσότερε προσπάθειε και να δαπανίσουμε ενέργεια και χρήμα προ αυτόν τον σκοπό. Επενδύσει λοιπόν χρειάζονται. Αυτό είναι ένα που πρέπει να κάνουμε. Ε, και κάτι άλλο είναι ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τον αποκλεισμό των νέων, μεγάλου αριθμού νέων, από την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Ζούμε σε κοινωνίες που βρίσκονται στην περιφέρεια και αντιμετωπίζουμε τεράστιε δυσκολίε ε, για να εντάξουμε του νέου στην κοινωνία. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλε περιοχέ τη Ευρώπη που βρίσκονται στην περιφέρεια τη Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με του νέου που είναι εκτό εκπαιδευτικού συστήματο ή επαγγελματική κατάρτιση ή ε, οποιοδήποτε εκπαιδευτικού συστήματο. Πρέπει να κάνουμε κάτι για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να είναι πιο φιλόδοξο και οι επενδύσεις που θα γίνουν να είναι καλές επενδύσεις για να δημιουργηθούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Τώρα, για τις πολιτικές, τις φορολογικές, ε, και τις οποίες θα χαρακτήριζα περισσότερο αναδιανομητικές παρά απλά ε, φορολογικές, θα πρέπει και αυτές να κατευθυνθούν προς τη δημιουργία θέσεων ε, Θέσουν εργασία για τους νέους σε περιοχές που υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες στην Ευρώπη. Επίσης, εσείς αναφερθήκατε στο κοινωνικό ισοζύγιο και για σας είναι κάτι σαν ένα μεγάλο καινούριο ευρωπαϊκό σχέδιο. Μακάρι. Και νομίζω πως η βάση για να το ε, ξεδιπλώσουμε αυτό το σχέδιο είναι το κείμενο του Κοινοβουλίου. Βέβαια έχουμε τον κοινωνικό πυλώνα που μέσω πρόθεσμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να καταπολεμήσει τις ανισότητες, αλλά και αυτό θα γίνει μέσω οικονομικών πολιτικών, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κοινωνικός πυλώνος έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όταν είναι κανείς Ευρωπαίος έχει μια ε, ελάχιστη τουλάχιστον αξιοπρέπεια προσωπική. Και μιλάμε για τους ίσους κανόνες παιχνιδιού για όλους, για το level playing field. Γιατί έχουμε ακούσει τι κάναμε στο παρελθόν, για τις διαφορές, για την έλλειψη συνοχής και όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν την αγορά εργασία. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα λυθούν από τη στιγμή που θα έχουμε κάποιε ελάχιστε κοινωνικέ βάσει, τι οποίε θα αποκτά κανεί απλώ και μόνο επειδή είναι Ευρωπαίο. Και πέραν αυτού, πιο πάνω από το ελάχιστο, ο καθένα ό,τι επιθυμεί. Αλλά να έχουμε αυτόν τον ελάχιστο κοινωνικό πυλώνα. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, τα εξή δύο για να έχουμε καλύτερη ενσωμάτωση, ε, για να έχουμε καταπολέμηση της ε, ανισότητας ε, κτλ. Πρώτον, Ευρωπαϊκή Ελληνική και μπορείτε να το ονομάσετε όπως θέλετε. Γιατί δεν μπορεί εμείς να δικαιολογούμε πως έχουμε ε, ταμεία για την άμυνα και ένα ταμείο για τις τράπεζες και τα καλωσορίζουμε, αλλά δεν έχουμε χρήματα για κανένα ταμείο έτσι ώστε να έχουμε τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο ενεργεία για όλους. Όχι. Πολιτικά αυτό δεν μπορεί να το πουλήσει κανείς και είναι και τελείως ανισόρροπο. Και κάτι που δεν θα αρέσει σε όλους, αλλά εμένα μου αρέσει να λέω αλήθειε, Η αρχή της επικουρικότητα δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί πρόφαση έτσι ώστε να επιτρέπουμε να συνεχίζουν ε, ζωντανές οι ανισότητες η Ευρώπη θα πρέπει να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν ανισότητες, τις βλέπει συνολικά και θα πρέπει να είναι ε, ενεργή έτσι ώστε να ξεπεραστούν. Τώρα υπάρχει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το basic income που λένε στα αγγλικά. Θέλουμε να το δούμε γιατί βήμα-βήμα το προσεγγύρινουμε και θα είναι δύσκολο να πετύχουμε το, το ελάχιστο ε, εγγυημένο εισόδημα γιατί είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο. Και ίσως είναι μία ιδέα για το μέλλον, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να το παγιώσουμε ως δικαίωμα για το άμεσο μέλλον στην Ευρώπη, πριν τη στιγμή που θα το εφαρμόσουμε και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρινακάρη. θέλει το λόγο. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για το γεγονός ότι ήρθατε στην συνεδρίασή μας και χαίρομαι που άκουσα ποια είναι τα σχέδιά σας. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε κάποια λόγια παραπάνω για τον κοινωνικό πυλώνα. Είναι ένα σημείο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ κοινωνικού πυλώνα και ευρωπαϊκού εξαμήνου. Γιατί κάποια από τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέσω του ευρωπαϊκού εξαμήνου έχουν αυξήσει την ανισότητα και έχουν δημιουργήσει προβλήματα, έχουν αυξήσει την παιδική φτώχεια, δυσκολέψει την εξέβρεση εργασία. Ξέρω πω προσπαθείτε μέσω του κοινωνικού πυλώνα να τα ξεπεράσουμε, αλλά μέσω αυτού του κοινωνικού πυλώνα θα υπερκεράσουμε τα όσα κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αν εκεί θεωρούμε ότι υπάρχει ε, κάποια διαφορά. Μα είπατε πω πρέπει να συνοδεύουν το ένα το άλλο. Φαίνεται λογικό αυτό, αλλά σε περίπτωση που υπάρχει αμφισημία μεταξύ τη κοινωνική διάσταση και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. ποιο κερδίζει τη μάχη αυτή. Και επίση θα ήθελα να μου πείτε Τι άλλο βρίσκεται στα σκαριά. Έχουμε άλλες νομοθετικέ προτάσεις. Μας είπατε πως έχετε μία που ετοιμάζετε. Για τον κοινωνικό πυλώνα λοιπόν έχουμε κάτι παραπάνω. Και το πρωτόκολλο που έχουν προτείνει τα συνδικάτα με τα δικαιώματα των εργαζομένων ε, που θα πρέπει ε, να κυριαρχούν ε, επί των δικαιωμάτων που έχει η νέα αγορά. Θα το δούμε αυτό κάπου. Το πιστεύει αυτό η Κομισιόν. Για την οικονομία του διαμοιρασμού και για τις πλατφόρμες, θα στείλετε και κάποιο έγγραφο για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτές τις πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού γιατί ξέρουμε ότι αρκετοί εργοδότες προσπαθούν να πείσουν που ότι είσαι ελεύθερος επαγγελματίας όταν εργάσαι για αυτούς και όχι εργαζόμενος με αποτέλεσμα να είναι διαφορετικά τα δικαιώματα τα οποία δικαιούσε. Οπότε για το θέμα αυτό έχετε κάτι ε, στο μυαλό σας. Κυρία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε που έχετε έρθει για να συζητήσουμε. Μας είπατε στην εισηγησία σας σήμερα το πρωί ότι πρέπει να έχουμε ελπίδα στο μέλλον της Ευρώπης. Διότι η πρώτη σα ομιλία σήμερα το πρωί, η εισηγησία σα ήταν βαθιά ανθρωπιστική και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα είμαστε μάρτυρε μια κρίσης στην ε, ουσία της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Εάν προσέχαμε όχι μόνο όλες οι πολιτικές μας να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά να ενημερώνουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες για το πόσο είναι σημαντικό να ανήκουν στην Ευρώπη, για το ότι η Ευρώπη τους ενώνει και ότι η Ευρώπη είναι το σύνολο των πολιτών της, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Εδώ λοιπόν θέλω να θέσω μια ερώτηση. Εργαζόμαστε σε πολλά επίπεδα και εργαζόμαστε εντατικά σε αυτή την Επιτροπή και μεταξύ των διαφορών επιτροπών για να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών διαστάσεων και των ε, οικονομικών προεκτάσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών. Όμω η πλειοψηφία αυτών των πολιτικών δεν φτάνουν στου Ευρωπαίου πολίτε, δεν του αγγίζουν. Και όταν του αγγίζουν, πολλέ φορέ δεν, τους, ε, δεν, δεν γίνεται κατανοητό. Αυτό καταλαβαίνω δεν είναι αποκλειστική ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ευθύνη πολλέ φορέ πάνω απ' όλα των ε, ίδιων των κυβερνήσεων των κρατών μελών όπως έλεγε ο Ντουράο Μπαρόζο, έχουμε την τάση να εθνικοποιούμε όλες τις ε, αρετές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξευρωπαίζουμε όλα τα προβλήματα. Ό,τι καλό ε, γίνεται το έχουν κάνει οι κυβερνήσεις και ό,τι πάει στραβά φταίνε Βρυξέλλες. Έτσι λοιπόν, κανεί δεν αναλαμβάνει στην ουσία ε, την ευθύνη τη πραγματικότητα. Ε, πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει ταυτόχρονα να πληροφορούμε του πολίτε για την κάθε μια από τι πολιτικέ που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε και η οποία ε, είναι στραμμένη και απευθύνεται στους ανθρώπους, στους πολίτες, ότι γίνεται για αυτούς. Λόγου χάρη τα κονδύλια της κοινή αγροτικής πολιτικής. Πρέπει οι αγρότες να καταλάβουν ότι η στήριξη που λάμβαναν δεν προερχόταν από τις εθνικές τους κυβερνήσεις, αλλά από το σύνολο των κρατών μελών. Το ίδιο η στήριξη προς τους ανέργους ή της ε, εκπαίδευσης των νέων. Ένας νέος όταν κάνει ένα στάζ, μια ε, μαθητεία, μια άσκηση, πρέπει να ξέρει ότι αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί αυτέ τι ευθύνε να τι εκχωρούμε στα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη-μέλη έχουν την τάση να ε, υπεξαιρούν κατά κάποιο τρόπο, να καταχρώνται τι θετικέ κινήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να οικοδομήσουμε σωστά την Ευρώπη. Ιδάλω θα παραμένουμε αποκλεισμένοι στι Βρυξέλλε ω ένα θεωρητικό ε, σχηματισμό, ένα οικοδόμημα που κανεί δεν ξέρει πολύ καλά σε τι χρησιμεύει. Και επίση ε, κάτι ακόμη για τα θέματα τη πληροφορία και τη ενημέρωση. Εδώ έχουμε μια Ευρώπη ε, μια Ευρώπη ξεχασμένη και παραγωνισμένη μεταξύ άλλων. Ε, πήγατε στην Πορτογαλία και είδατε τι γίνεται με τις δασικές πυρκαγιές. 74 τουλάχιστον έχασαν τη ζωή τους και 50 ε, είναι τραυματίες. Ε, σας ευχαριστώ για τα λόγια που είπατε στην Πορτογαλία και τα συλληπιτήρια που εκφράσατε, όμως πρέπει να σκεφτούμε και τους ανθρώπους της υπαίθρου τι εκπροσωπεί αυτή η περιοχή τη Ευρώπη. Όταν θα ετοιμάσουμε το επόμενο, όταν θα σχεδιάσουμε το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι πολιτικέ μα, όλε τι γραφικέ περιοχέ, θα απευθύνονται και σε αυτού του ανθρώπου. Ότι οι εθνικέ κυβερνήσει, όταν με τη σειρά του σχεδιάζουν τα δικά του επιχειρησιακά προγράμματα, θα λάβουν μέρημνα για του ανθρώπου αυτού. Θα βεβαιωθούν ότι τα χρήματα αυτά πάνε στα χέρια αυτών των ανθρώπων, ότι τα κονδύλια φτάνουν στι περιοχέ τη υπαίθρου που είναι πιο αποκλεισμένε, που βρίσκονται σε περιοχέ απομακρυσμένε, σε εξόχου απόκεντρε περιοχέ. Αυτό πρέπει να γίνει διδάλωση, οι ανισότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνουν ω έχουν. Και για τι πολιτικέ τη συνοχή. Πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Εδώ πραγματικά απευθύνω μια ισχυρή έκκληση στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να μα βοηθήσει να έχουμε διαρκώ κατά νου ότι θέλουμε Ευρώπη των πολιτών. Αλλά δεν θα την έχουμε εάν δεν έχουμε πολιτικέ που ε, λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες αυτών των πολιτών και ταυτόχρονα ε, ε, διαμορφώνουν από κοινού την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή. Ευχαριστούμε, ο Χάβι Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα όσα μας εξήγησε, για το όραμα το οποίο μοιράστηκε μαζί μας και με το οποίο θα συνταχθώ σε μεγάλο βαθμό. Χρειάζεται η Ευρώπη μια ευκαιρία για να αναδιοργανωθεί μετά τα τόσο δύσκολα που πέρασε πέρσι, για να ξαναβρει τον εαυτό της. Και δεν είναι μόνο ευκαιρία αυτό, αλλά και τεράστια ευθύνη, ε, γιατί κάποιες από τις ιδέες τις οποίες εμείς εκπροσωπούμε στον κόσμο, που είναι ο το κοινωνικό μοντέλο της αγοράς, το ότι θα πρέπει η παγκοσμιοποίηση να ακολουθεί κανόνες, να έχουμε μια διανομή των κερδών της, ή θα τις υπερασπιστούμε εμείς ή δεν υπάρχει άλλος. Άρα λοιπόν και ευκαιρία και ευθύνη. Και πρέπει να δώσουμε και μία απόκριση στους ε, Ευρωπαίους πολίτες και να τους ρωτήσουμε καταρχήν τι επιθυμούν. Θέλω μια Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω, πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική, γιατί δυστυχή τα τελευταία χρόνια δεν ήμασταν σε κοινωνικό επίπεδο αποτελεσματικοί, ενώ στο παρελθόν ήταν ένας μηχανισμός πάρα πολύ αποδοτικός, γιατί ούτε οικονομικά ήμασταν αποτελεσματικοί με τις δυσλειτουργίες που ήταν πολλές και πρέπει να το δούμε αυτό μέσα στο ενίο νόμισμα και όχι μόνο και με άλλες ε, κρίσεις που περάσαμε, χρειάζονται μια πιο δίκαιη Ευρώπη, Κάτι το οποίο και αυτό έχει τονιστεί και όταν λέμε πιο δίκαιη είναι γιατί η ανισότητα δημιουργεί, μάλλον διαβρώνει την ε, αξιοπιστία των θεσμών. Και εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που μας οδήγησαν σε αυτό που συμβαίνει σε πολλά άλλα σημεία του δυτικού κόσμου. Δηλαδή θα πρέπει να αποκριθούμε σε αυτές τις ανησυχίες και κυρίως ανησυχίες που προκαλεί παγκοσμιοποίηση και το ξέρετε, το είπατε, με μηχανισμούς που σε εσωτερικό επίπεδο θα φέρουν κάποιο είδους αντίβαρο και θα προετοιμάσουν τους ε, συμπολίτες μας για να γίνουν πιο ε, δυνατοί και εντός και εκτός και να επηρεάζουμε περισσότερο τα πράγματα. Εμείς έχουμε πολλές προτάσεις στη δική μας ομάδα, τις οποίες στους τελευταίους μήνες καταθέτουμε. Καταρχήν, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Πυλώνας. Ξέρω πως εσείς στην Κομισιόν δίνετε μεγάλη σημασία και το ζήτημα είναι πώς αυτός ο κατάλογος αγαθών προθέσεων μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματική επιβολή από πλευρά κρατών μελών, να προσγειωθούμε δηλαδή στην πραγματικότητα, γιατί με το να μοιραζόμαστε αυτό το πλαίσιο αναφοράς που είναι ο κοινωνικός πυλώνας και που περιγράφει αυτός, χρειαζόμαστε τα ισχυρά νομικά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να εφαρμοστούν όλα αυτά και στην πράξη. Εμείς βάλαμε λοιπόν στο τραπέζι την ανάγκη να έχουμε για παράδειγμα μία οδηγία για τις ε, συνθήκες εργασίας. Ξέρετε πως έχουμε τέτοιες μεταλλάξεις στην αγορά εργασίας οι οποίες δημιουργούν πάρα πολλές από αυτές τις ανησυχίες από τις οποίες πλήττονται οι Ευρωπαίοι. Δεύτερον, η εγγύηση για τα παιδιά. Και αυτή τη στιγμή είναι και πιλωτικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η παιδική φτώχεια είναι ένα από του μεγάλου κινδύνου που αντιμετωπίζουμε. Θεωρούμε πω είναι μια πολύ καλή ιδέα και θα πρέπει να την προωθήσουμε. Τρίτον, πώ θα δώσουμε μια νέα ισορροπία μεταξύ Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και κυρίω του κομματιού που είναι το πιο σκληροπυρονικό, σκληροπυρονικό σε μακροοικονομικά θέματα, που έχει μεγάλη δυνατότητα επιβολής, πώς αυτό λοιπόν μπορούμε να το επαναπροσδιορίσουμε και να το εξισορροπήσουμε με αυτήν την κοινωνική διάσταση που επιδιώκουμε. Και το κάνετε αυτό την αρχή της θητείας σας και τώρα έχουμε αρχίσει να το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Οπότε πώς θα κάνουμε αυτόν τον επαναπροσδιορισμό έτσι ώστε το πιο σκληρό κομμάτι να το απαλύνουμε. Τι γίνεται με τη φτώχεια, με την ανισότητα, με, την με τον κοινωνικό ε, αποκλεισμό. Οι ιδέες είναι πολλές και θετικές. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ταμείο για την ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλά έχουν συζητηθεί. Εμείς προτείναμε μία πράσινη βίβλο για την ε, ανισότητα στην Ευρώπη. Οι προτάσει είναι πολλέ και καλέ. και στα δύο χρόνια που μένουν, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, τόσο μαζμένοι, πώς θα μπορέσουμε αυτό να βάλουμε πραγματικά στα σκαριά κάποιε από αυτέ τι καλές προτάσεις που είναι στο τραπέζι, διαφορετικά αυτό θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο για το μέλλον τη Ευρώπη. Έχω δύο ακόμα ονόματα στον κατάλογο. Θέλετε να του ακούσετε και μετά να απαντήσετε. Πολύ ωραία. Η κυρία Κούνεβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ότι ήρθατε σήμερα να συζητήσετε όλοι μαζί μας. Και στο πλαίσιο της συζήτησης για την προετοιμασία του Μελλοντικού Προγράμματος Εργασίας της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και επειδή εσείς τονίσατε την μεγάλη σημασία της απασχόλησης, θα ήθελα να θέσω απόψη μια πρωτοβουλία την οποία έχουν αναλάβει κάποιοι υπουργοί στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Ελληνίδα αναπληρώτρια υπουργό εργασία μαζί με άλλου συνάδελφου τη στηρίζουν μια πρόταση σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες που τα προορίζονται για προγράμματα απασχόλησης και τα, τα χρηματοδοτούνται είτε από κοινωνικούς ή από άλλους πόρους θα έπρεπε να εξαιρούνται από το υπολογισμό του ελλείμματος σύμφωνα με το σύμφωνο σταθερότητας. Με τον τρόπο αυτό θα τονωθεί η εργασία η οποία υποφέρει από τα μέτρα λιτότητας, θα δώσουμε σανίδα σωτηρία στους ανθρώπους και θα στηρίξουμε την αξιοπιστία της Ευρώπης. Επίσης, αναρωτιέμαι αν έχετε σκεφτεί τι μπορεί να γίνει, πώς να οργανώσουμε έτσι την Ευρώπη, ώστε να βγάζουμε τους μεσάζοντες που κρατάνε τις θέσεις εργασίας και μοιράζονται ανά έξι μήνες εργασία σε κάθε εργαζόμενο. Αυτή η χρήση έχει απλωθεί και αυξάνει την ανισότητα στην Ευρώπη, τον διχασμό στην κοινωνία μας και τη φτώχεια. Νομίζω έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μπροστά μας και όλο και περισσότερο αυξάνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε η εργασία να είναι άμεση για το εργαζόμενο, όχι μέσα από μεσάζοντες. Θα στηρίξετε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς ως Επίτροπος Αρμόδιος για τις θέσεις εργασίας με τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος... Ο κύριος Χότς. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω που οργανώσατε αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων και ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν που ήρθε εδώ. Η αρχική γενική μου παρατήρηση είναι ότι τα λόγια σας ήταν όμορφα. Αυτά που είπατε ακούγονται πολύ ωραία, Αντιπρόεδρε. Οι εξωτερικές και εσωτερικές δυσχέρειες θα πρέπει να μας ε, κάνουν να είμαστε πιο ενωμένοι, να συσπηρωθούμε και να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μια ένωση αξιών. Πρέπει να περάσουμε από την περίοδο τη κρίση ε, στην ανοικοδόμηση ενό νέου μέλλοντο. Είναι πολύ όμορφα λόγια αυτά, όμω δεν μεταφράζονται νομίζω σε καθημερινή εμπειρία, στην, ε, στο τι συμβαίνει στην καθημερινότητα και σε πράξει. Δεν στηρίζονται αρκετά από την κατάλληλη δράση. Άρα μπορεί να είναι πολύ ωραία ρητορικά σχήματα αυτά που είπατε, αλλά Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Αντιπρόεδρε. Αυτές οι εξωτερικές προκλήσεις σας φέρετε να ενοποιούν την Ευρώπη, λόγω χάρη οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις μετακατάστασης για τις πρόσφυγες ή οι οδηγίες για τις μεταφορές. Ε, η μετατροπή του πολωνικού ε, στόλου μεταφορών στις οδικές μεταφορές, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη. Ε, Πώς θα ενισχυθούμε από αυτά που προτείνεται. Μετά οι με μέτρων για την ενέργεια, η οδηγία για τα λοιπάσματα. Αυτά αποσταθεροποιούν την γεωργία μα και τι εταιρείε και επιχειρήσει μα. Ή για την κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχουν ακόμα σοβαρέ ανισότητε στι άμεσε επιδοτήσει. Ιδίω τι χαμηλότερε για του γεωργού από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Το Nord Stream 2 αυτός ο αγωγός μας ενώνει, αυτές οι εξωτερικές προκλήσεις μας ενώνουν. Ή ε, μήπως τελικά το αντίθετο συμβαίνει, μήπως απέναντίας μας χωρίζουν, μήπως δημιουργούν αφορμές για να χωριστούμε περισσότερο. Ε, Βαριετάτε κονκόρντια είναι υποτίθεται το σύνθημά μας, ενωμένη στην ποικιλομορφία. Όμως, Θέλουμε να το δούμε και στην πράξη. Και κατά δεύτερον, όταν μιλάτε για τον κοινωνικό πυλώνα, πρέπει να έχουμε διαρκώς κατά νου και να θυμόμαστε ότι βάζει τις αρχές της επικουρικότητας αυτοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές είναι τα κράτη-μέλη. Άρα ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορούν να στηρίξουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, μπορούν να στηρίξουν τους εργαζομένους και τους νόμους περιεργασίας. Προφανώς το χρειαζόμαστε και αυτό για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εάν παρέμβουμε υπερβολικά, θα γίνει ανταπαραγωγική η παρέμβασή μας. Γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι συγκρατημένες και ισόρροπες. Η ευρωπαϊκή ένταξη και η κοινωνική πρόοδος, όπως τόσο ωραία το είπατε, ναι, αλλά με τρόπο ισόρροπο. Και τελευταίο σημείο, πολύ σύντομα, η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση βεβαίω και σημαίνει ωφέλη, όμω σημαίνει και δυσκολίε, δυσχέρειε και απειλέ. Ε, για να το πω ξεκάθαρα, στην ε, παγκοσμιοποίηση που σήμερα διαμορφώνεται, βλέπουμε πολύ συχνά κερδισμένου και ιτημένου. Οι κερδισμένοι παίρνουν όλα τα ωφέλη και οι ιτημένοι είναι αυτοί που ε, γνωρίζουν την δικτατορία και την ποδηγέτηση στις επιχειρήσεις και τις εταιρείε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει προβλήματα και στο κοινωνικό τη ιστό. Δεν έχουμε πραγματική ισότητα και μόνο οι πιο ισχυροί φαίνεται ότι θα επιβιώσουν. Όλα αυτά λοιπόν τα ωραία λόγια καλό είναι να μεταφράζονται και σε πραγματικές χειροπιαστές πράξεις οι οποίε πραγματικά θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια ολοκληρωμένη Ευρώπη και να ενωθούμε. Όμως δεν θα επιτρέψουμε η Ευρώπη να γίνει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χότ. Τώρα να δώσω τον λόγο και πάλι στον Αντιπρόεδρο. Πολλές οι ερωτήσεις, αλλά ε, πιστεύω ότι θα μπορέσετε να τις απαντήσετε τέλεια όλες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις και φοβούμαι ότι δεν μπορώ να δώσω διεξοδικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Ενδεχομένως η συνάδελφος Τάισεν να απαντήσει σε κάποιες άλλες από τις ερωτήσεις σας. Αλλά θα προσπαθήσω. Θα ξεκινήσω από την παγκοσμιοποίηση. Η γενική αίσθηση σε κάποιες χώρες, όχι σε όλες, σε κάποιες, είναι ότι η παγκοσμιοποίηση αυτή καθεαυτή ε, προξενεί αυτό το, την αίσθηση ότι υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Δεν είναι έτσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια χώρα που έχει χαρακτηριστεί και υπόδειγμα για την κοινωνική της πρόνοια σε όλο τον κόσμο, τη Σουηδία. Ο λόγος που η Σουηδία έχει μια τόσο γενναιόδορη κοινωνική πρόνοια είναι επειδή παίρνει χρήματα εκτός της δικής της οικονομίας. Είναι ένα άριστο παράδειγμα όπου εξωτερική ανταγωνιστικότητα, κοινωνική ένταξη και κοινωνική πρόνοια έχουν μπει στο ίδιο σακούλι, χωρίς την κοινωνική πρόνοια και την ε, κοινωνική ένταξη και μια τέτοια διάθεση συμμετοχικότητα στη σουηδική κοινωνία, η Σουηδία δεν θα ήταν ανταγωνιστική προς τα έξω. Και αν ε, αυτή η χώρα δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική, οι εταιρείε τη αυτέ δηλαδή που μπορούν να κινηθούν και στο εξωτερικό δεν θα έπαιρναν τόσο καλέ συμφωνίε, δεν θα πετύχαιναν τόσο καλού όρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπει χρήμα και να χρηματοδοτηθεί η κοινωνική πρόνοια τη χώρα. Αυτό ε, το παράδειγμα για μένα είναι μια απτή απόδειξη ότι η παγκοσμιοποίηση δεν προκαλεί αναγκαστικά ε, διέρεση και διχασμό στα κράτη. Όλα εξαρτώνται από το πώς αξιοποιούν τα κράτη-μέλη το εισόδημα που παίρνουν από την παγκοσμιοποίηση. Η Σουηδία είναι τελείω ανοιχτή ε, στην ε, παγκοσμιοποίηση. Αλλά έχει και μια από τι καλύτερε κοινωνικέ πρόνοιες και κοινωνική προστασία. Υπάρχει ένας σαφέστατος συσχετισμό μεταξύ των δύο. Γι' αυτό Ελπίζω οι πολιτικοί να αρχίσουν να επικεντρώνονται σε πραγματικά γεγονότα και όχι να κατηγορούν την ανοιχτή παγκοσμιοποίηση, την ανοιχτή οικονομία. Η δομή των κοινωνιών μα είναι ένα πρόβλημα, όχι η ανταγωνιστικότητα. Αυτό δημιουργεί πραγματικά προβλήματα. Βεβαίω είναι εξίσου αληθέ ότι κάποιοι στην παγκοσμιοποίηση δεν θα τα βγάλουν πέρα γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν στην αγορά. Εκεί δεν μπορούμε να επιδοτήσουμε μια ακατάλληλη παραγωγή. Πρέπει να κοιτάξουμε τις επενδύσει για το μέλλον, λόγου χάρη. Είναι ένας διαρκής, ε, μια διαρκή σχέση ανταγωνιστική, μια διαρκής εξέλιξη αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ο ρόλος της κοινωνικής πρόνοιας είναι να αυξήσει την αντοχή, την ανθεκτικότητα. Και ο στόχος της ανθεκτικότητα είναι ακριβώς οι άνθρωποι να μπορούν να προσαρμόζονται, να είναι πιο δημιουργικοί, πιο επινοητικοί, να είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Και όχι απλώς να το υπομένουν, όχι απλώς να είναι αποδέκτες των εξωτερικών πιέσεων. Άρα, το να μετακινηθούμε από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει τώρα η κοινωνία. Θέλουμε μια κοινωνία δυναμική. Μια κοινωνία που να είναι σε θέση να αντιδράσει και να διαμορφώσει το δικό της μέλλον, το πάρει στα χέρια της. Το κατά πόσον είμαστε ενωμένοι ή όχι. Φυσικά και υπάρχουν ε, διαφωνίες μεταξύ των ε, πολιτικών κομμάτων και μεταξύ των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι είμαστε τώρα περισσότερο ενωμένοι από ποτέ. Υπάρχουν ζητήματα όπως οι ποσοστώσεις ε, των προσφύγων. Ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει αυτή την πρόταση είναι ότι βασιζόμαστε σε αξίες. Εάν ε, λέμε ότι θέλουμε να φροντίζουμε ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινα όντα, είναι δίκαιο και επιβάλλεται να κατανεμηθούν οι ευθύνε. Βασιζόμαστε σε αξίες υποτίθεται. Το ίδιο και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι ζωτική σημασία. Δυστυχώς, Έχουμε περάσει σε μια περίοδο που εγώ τουλάχιστον προσωπικώς δεν πίστευα ότι θα ξαναβιώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ε, αμφισβητούμε πράγματα τα οποία θεωρούνταν δεδομένα. Εγώ νομίζω ότι οι αυτοί είχαν περάσει στην Ευρώπη. Και όμως έχουμε το χωρίσει. Αυτό είναι πολύ καυτό θέμα. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα αυτά ε, και να τα αντιμετωπίσουμε θαραλέα. Διότι αν δεν πιστεύουμε στο κράτος δικαίου, δεν έχουμε τίποτα. Η Ένωση είναι Ένωση κράτους δικαίου. Οι αξίες της Ένωσης ε, βασίζονται σε αυτό. Ακόμη και αν κάποιοι λένε ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, ερμηνείες του κράτους δικαίου, ε, δεν μιλάμε και για πυρηνική φυσική. Έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να ε, αναλύσουμε, να εξετήσουμε σωστά τα συστήματά μας και υπάρχουν συστάσεις προς τα κατημέλια για να ε, μπορέσουν ε, να ε, προωθήσουν το κάτω δικαίου και να αναλάβουν τις σωστέ πρωτοβουλίες Για την ανεργία των νέων, την αγγίση των νέων και τον συνδυασμό των δεξιοτήτων με την διαβίωμάθηση. Είναι αλήθεια ότι η εγγύηση των, νέων πρωτοβουλία αυτή σε κάποιε περιπτώσει τα έχει πάει καλά, σε κάποιε άλλε λιγότερο. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέραν του να προβλέπει και να στοχεύει πόρου είναι να συνεργαζόμαστε στενότερα με τα κράτη-μέλη ώστε να υλοποιήσουν σωστά και να μάθουν από του άλλου. Να δουν δηλαδή ποιε είναι οι καλέ πρακτικέ για να υπάρξει καλύτερη υλοποίηση. Και στι πολιτικέ τη απασχόληση και στην εγγύηση των νέων. Ε, υπάρχουν ε, κριτικά, επικριτικά σχόλια, τα οποία είναι και εύστοχα. Γι' αυτό προσπαθούμε να ξαναδούμε αυτές τις πολιτικές και να μάθουμε από το τι έχει συμβεί ως τώρα με αυτές για να υλοποιήσουν καλύτερα και την εγγύηση των νέων ε, οι χώρες. Σε κάποια πράγματα τα έχουν πάει καλά οι χώρες. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλλον τα έχουν πάει καλά οι χώρε, όπως η Ισπανία. Ο Ισπανό συνάδελφος εδώ είπε και έχουμε δει η εγγύηση των νέων να φέρνει και κάποιε αναγκαστικέ μετατροπέ στην πολιτική απασχόληση και την πολιτική για του νέου. Οι νέοι έχουν ωφεληθεί από αυτά. Έχουν ωφεληθεί από την ε, εργατική πολιτική. Ίσως να μην φτάνει αυτό, ίσως οι μετατροπές να μην ήταν τεράστιες, όμως ήταν ήδη κάτι. Και σχετίζονταν όλα αυτά με την εγγύηση για τους νέους. Η ποιότητα λοιπόν είναι ακόμη πιο σημαντική από το ίδιο το ποσό, το χρηματικό ποσό. διότι δεν αρκεί κανείς ε, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα να ε, χρησιμοποιήσει απλώς περισσότερο, όταν ένα μάξι δεν ε, προχωράει, δεν αρκεί να του φορτώσεις περισσότερη βενζίνη. Ούτε μετράει το ποσό πρόσφατα πριν γέμισε τον το τεπόζιτο. Έτσι λοιπόν τα κάτι μέλη κάνουν ό,τι μπορούν και με αυτό το θέμα. Μπορούν να το έχετε ακούσει πολλές φορές και προηγουμένω από μένα, αλλά αν ήμουν δικτάτορα τη Ευρώπη, το πρώτο που θα έκανα θα ήταν να ε, μεταρρυθμίσω τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών, ώστε να έχουν τα αποτελέσματα των καλύτερων της Ευρώπης όλοι. Αυτό είναι το κλειδί για όλα. Είναι σημαντικό για τους νέους, είναι σημαντικό για την αντιμετώπιση της ενεργείας των νέων και είναι και σημαντικό από την άποψη της κοινωνικής δικαιοσύνης επίσης. Εάν δούμε και τις περιοχές της Υπέθρου που έφυξε η κυρία Ριμπέρου, υπάρχουν τομεακές πολιτικές για τις περιοχές της Υπέθρου, όμως μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των, των ανθρώπων των περιοχών της υπαίθρου, εάν οι οριζόντιες οι οριζόντιε πολιτικέ μα, λόγω χάρη οι εκπαιδευτικέ πολιτικές, υπάρχουν χώρες και γεωγραφικές περιοχές όπου η ποιότητα τη εκπαίδευση είναι χειρότερη στις περιοχέ τη υπαίθρου από ό,τι στι αστικέ. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος οι ίδιοι δάσκαλοι που έχουν την ίδια εκπαίδευση και κατάρτιση και υποτίθεται ότι είναι έτοιμοι να διδάξουν. Είναι έτοιμοι να προσφέρουν την ε, υπηρεσία τη ίδια ποιότητα στα παιδιά να μην το κάνουν. Δυστυχώ δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η δική μου αποστολή ω επιτρόπου, ή τέλο πάντων μία από τι βασικέ μου αποστολέ, είναι να φέρω ε, να συμπεριληφθούν τα θέματα του εκπαιδευτικού συστήματος και της παιδείας στις αναχώρα συστάσεις. Θέλω να επικεντρωθούμε περισσότερο στα εκπαιδευτικά συστήματα και την εκπαίδευση των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, των ίδιων. Είναι πολλές οι χώρες όπου αυτές οι δυσκολίες είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικές. Καμιά φορά οι προσπάθειες για αλλαγέ φαίνεται να είναι ε, χαμένες στην αιωνιότητα. Χρειάζονται πολλά χρόνια για να γίνει πραγματικότητα μια αλλαγή. Αλλά δείτε τι έγινε στην Εστονία και την Πορτογαλία λόγω χάρη. Μιλάμε για δύο χώρες που κατάφεραν να βελτιώσουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Δείτε λόγω χάρη τη μελέτη του ΟΣΑ, ε, του, της πίζας, ε, για το σύστημα της πίζας και για την Πορτογαλία και την Εστονία. Η Πορτογαλία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε χάρη στις μεταρρυθμίσεις της να προχωρήσει πάρα πολύ ε, στους δείκτες της πίζας. Άρα Ακόμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να πετύχουμε πολλά, ακόμα και αν χρειάζονται πολύ περισσότερα μακροπρόθεσμα. Αν κανεί στραφεί και αντιμετωπίσει τα σωστά προβλήματα. Αυτό είναι πραγματικά στην καρδιά όλων των ζητημάτων για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την ανταγωνιστικότητα. Και είναι ακόμη πιο σημαντικό όταν πρέπει να, προσαρμοστούν, ε, να προσαρμοστούμε και καλούμαστε να προσαρμοστούμε στην ψηφιακή εποχή. Λίγα λόγια τώρα για το κοινωνικό πυλώνα και το εξάμεινο. Όπως ξέρετε, ο ρόλος του κοινωνικού πυλώνα είναι να θέσει τις αρχές για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ε, ισότιμη αγορά εργασίας και την ισότητα. Αυτές οι αρχές αντικατοπτρίζονται και στις ε, διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται οι διάφορες χώρες. Δεν υπάρχει μία λύση που να είναι ίδια για όλους. Υπάρχουν διαφορές στην οικονομία των χωρών μεταξύ τους, στις αγορές εργασίες, στο τι συμβαίνει στον κάθε κλάδο και τομέα, στη φορολογία. Είναι πολύ διαφορετικά όλα αυτά. Οι πρακτικές ε, για την ε, αγορά εργασίας και την πολιτική τους ή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Παρ' όλα αυτά θελήσαμε να ορίσουμε κάποιες βασικές αρχέ τι οποίες να μπορούμε να ακολουθήσουμε ε, κατά τη διάρκεια τη διαδικασία του εξαμήνου. Κυρία Καρή, θέσατε το εξή θέμα. Κάποιες φορές ο κοινωνικός πυλώνας μπορεί να συμπληρώνει το ευρωπαϊκό εξάμεινο να επικαλύπτονται αυτά τα δύο. Ε, μπορεί να συμβεί αυτό, πάντοτε συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Η αναχώρα κάποιε κάποιες φορές, ορισμένα σημεία τους ε, έχουν πιο σοβαρές συστάσει από ότι κάποια άλλα. Όμως και πάλι θέλω να δώσω εδώ ω παράδειγμα την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία βρισκόταν σε δυσχερέστατη οικονομική θέση και ταυτόχρονα έδειξε ότι μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευσή τη, που τώρα ήδη δίνουν του πρώτου καρπούς. Ε, δεν είχαμε τότε τον κοινωνικό πυλώνα όπως βρίσκεται σήμερα, Όμω, εάν θελήσει κανεί να επικεντρωθεί στην ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ε, ένταξη και την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών τον οποίων μέρος είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και η παιδεία, ε, αυτά δεν αντιφάσκουν αναγκαστικά με μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική λόγου χάρη και τις ε, συγκεκριμένες δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν προδιετίας λόγου χάρη. Το νομικό καθεστώς του κοινωνικού πυλώνα Στη φάση αυτή είναι ένα σύνολο από αρχέ που μπορεί να μεταφραστούν σε συγκεκριμένε δράσει κατά τη διάρκεια τη διαδικασία του εξαμήνου και με μακροπρόθεσμα θα πρέπει να οδηγήσουν σε αναχώρα συστάσει. Για την κυκλική οικονομία και τη συμμετοχική οικονομία δεν βρίσκω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, καθότι στον τομέα αυτό Όλοι θα πρέπει να σέβονται τα ίδια εργατικά δικαιώματα και τι υποχρεώσει που εκπληγάζουν από το δίκαιο. Ε, στην συμμετοχική οικονομία τα πράγματα ίσω να είναι λίγο διαφορετικά. Ε, εδώ λοιπόν, ε, πριν από λίγο καιρό, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε πώς μπορεί να είναι ε, τα πράγματα για έναν επιχειρηματία. Εάν συγκρίνεται λόγω χάρη το Airbnb με το Uber, αυτά χρησιμοποιούν ε, πλατφόρμες στο ίντερνετ. Κάποιο που νοικιάζει το διαμέρισμά του σε έναν άλλο ιδιώτη. Είναι επιχειρηματία, ε, είναι εργαζόμενος Και πώ μπορεί να συγκριθεί με αυτόν που εργάζεται για το Uber. Η οικονομία λοιπόν διαμερισμού, η συμμετοχική οικονομία διαμοιρασμού, ε, η οικονομία αυτή που επιτρέπει τη συμμετοχή όλων ε, είναι κάτι που πρέπει να δούμε πώς θα διευθετηθεί. για τον ελάχιστο μισθό. Ε, ο ελάχιστο μισθό πρέπει κάπω να συνδυάζεται και με κοινωνικέ υπηρεσίε και την κοινωνική ασφάλιση. Ο συνδυασμό αυτό διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε ελάχιστο μισθό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά το ελάχιστο εισόδημα έχει προκύψει ως προβληματισμός στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Έχουμε λοιπόν εντοπίσει 10 χώρες φέτος όπου έχει τεθεί το θέμα του ελάχιστου εισοδήματο. Και έχει προταθεί στα κράτη-μέλη να κοιτάξουν τι θα κάνουν με το πρόβλημα αυτό, γιατί υπάρχει θέμα διαφορετικό, υπάρχει θέμα ανισότητας. Κάποιες φορές ε, διαφέρουν άλλα πράγματα όπως ε, τα επιδόματα ανεργίας ή άλλες εγγύησεις που προσφέρουν τα κοινωνικά συστήματα αλλά η Επιτροπή κοιτάζει το ελάχιστο εισόδημα ως ένα θέμα που είναι πολύ πιο επίκαιρο από ό,τι προηγουμένω και προσπαθούμε να εντοπίσουμε διαφθορτικά προβλήματα στα επιμέρους για να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι. περνάει και ο χρόνος. Η κυρία Κούνεβα είπε ότι οι κοινωνικές δαπάνες και εάν αυτά που γίνονται για τις κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να αποκλείονται από το να μην υπολογίζονται στο μοσονομικό σύμφωνο, στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Πρόσφατα συζητήσαμε τον χρυσό κανόνα. Παραδοσιακά η ιδέα αυτή συζητιόταν στο επίπεδο των επενδύσεων. Εάν οι δαπάνε για τι επενδύσει θα πρέπει να αφαιρούνται από τα όσα προβλέπει το σύμφωνο. Έχουν γίνει κάποιε συζητήσει, ιδίω πριν από ένα-δύο χρόνια, για το αν οι στρατιωτικέ, οι δαπάνε θα πρέπει να περιλαμβάνονται ή όχι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλες οι δαπάνες θα έπρεπε να είναι στα κρατικά βιβλία. Αν υπάρχει έλλειμμα, υπάρχει έλλειμμα, ό,τι και αν θέλει κανείς να αφαιρέσει από το σύμφωνο. Να το εξηγήσω. Εάν αποκλείσουμε όλες τις κοινωνικές, αν αφαιρέσουμε όλες τις κοινωνικές δαπάνες, 60% του προπολογισμού στα περισσότερα κατημέλη, μένει 40% των δαπανών για να υπολογιστούν και στο σύμφωνο. Εάν περιορίσουμε το πεδίο μόνο στην απασχόληση, προκύπτει το εξή ερώτημα. Τι πρέπει να υπολογιστεί σε αυτό το σύνολο. Το πιο προφανές τμήμα των δαπανών είναι οι πολιτικές απασχόλησης. Αλλά τι θα κάνουμε με την εκπαιδευτική πολιτική. Όλη την ε, πολιτική παιδεία ή ένα μέρος της θα υπολογίσουμε ας πούμε. Τι να κάνουμε με τα προγράμματα επιδομάτων ανεργίας ή τις επενδύσεις. Αρχίζει και γίνεται πολύ δύσκολο δηλαδή. Δεν ε, λέω ότι είμαι καταρχήν αντίθετος λόγω των τεχνικών δυσκολιών, αλλά όταν μιλάμε για κοινωνικές δυσκολίες και προκλήσεις και προβλήματα απασχόλησης, Πρέπει να έχουμε και υγιή δημοσιονομικά. Είναι προϋπόθεση για την καλή απασχόληση και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης μακροπρόθεσμα. Τι άλλο. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα. Α, ένα ακόμα σημείο. Να έρθω πάλι στον ε, χώρο της εκπαίδευσης και της παιδείας. Μερικές φορές Είναι ευχάριστο να βλέπουμε ότι ακόμη και ένας επίτροπος μπορεί να περάσει τις ιδέες του. Ε, ξεκίνησα μια ιδέα που πριν από δύο εβδομάδες συμπεριελήφθη σε ε, μια ανακοίνωση για την ε, πολιτική παιδεία που πρόκειται σύντομα να δημοσιευτεί. Θα είναι μια εθελοντική ομάδα δράσης των κρατών μελών που θα θέλουν να μεταρρυθμίσουν τα εκπαιδευτικά του συστήματα. Και η ιδέα εδώ είναι να συγκεντρώσουμε τα κράτη-μέλη που θέλουν να βελτιώσουν λίγο χάρη την ποιότητα τη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι υπηρεσίε του ΩΣΑ και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να προσφέρουν τεχνική συνδρομή στα κράτη-μέλη. Να του δείξουν πού μπορούν να κάνουν τι σωστέ κινήσει και να αναλύσουν τι πρέπει να γίνει, χρησιμοποιώντα τι βέλτιστε πρακτικέ που ήδη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τώρα θα γίνει μέρος της εργαλειοθήκης μας. Εάν ε, σας ε, ε, αφορούν όλα αυτά, να φροντίσετε να μεταφέρετε το μήνυμα στις κυβερνήσεις σας. Υπάρχει και αυτό το εργαλείο τώρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος ή η διαβημάτιση ή η διαβημαθηση η η εκπαιδευση των εκπαιδευτικών. Είναι πολύ σημαντικό για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών στις κοινωνίες μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και να σας ευχηθώ πολύ καλό μεσοκαλό καιρό. Μεγάλο θέμα για τις σκανδιναβικές χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα τι είπες στην εισαγωγή σου και θα ήθελα κι εγώ να τονίσω πως πρέπει να δημιουργήσουμε τους νέους 27. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μετά το Brexit σαν να μην έχει γίνει τίποτα και νομίζω ότι είναι, αυτό είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας, για όσους θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή ε, Ένωση καινούρια. Σας ευχαριστώ που μας διαθέσατε τόσο χρόνο και που μας κάνατε πολλές ερωτήσεις και μας δώσατε και πάρα πολλές απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ.